χρόνο. Θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο έτσι κι αλλιώ για να απαντήσει σε μια προφορική ερώτηση που τη γνωρίζει σίγουρα αλλά που δεν θα παρουσιαστεί προφορικά. Έχετε το λόγο κύριε Επίτροπε. Yes, indeed, Mr. President, uh, members of... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές. Η Κομισιόν αποδίδει μεγάλη σημασία στην ε, ασφάλεια και την υγεία ε, στο χώρο εργασίας ε, και είναι πολλές οι πρόοδοι που έχουν σημειωθεί σε αυτό το τομέα. Η στρατηγική της Ένωσης από το 2007 μέχρι το 2012 είχε θετικό αντίκτυπο σε ολόκληρη την Ένωση ε, και αυτό το επιβεβαιώνει και η αξιολόγηση που έγινε, η οποία δεν επιβεβαιώνει και την ευρωπαϊκή διάσταση της πολιτικής αυτής και της στρατηγικής προσέγγισης μας. Και αυτή ήταν ιδιαίτερα σκόπιμο όσον αφορά το θετική τάση, όσον αφορά τη μείωση των εργατικών ατυχημάτων και τη βελτίωση της εφαρμογής της ε, νομοθεσίας σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας. Επιβεβαιώνει δε ότι 25% μείωση των εργατικών ατυχημάτων θα είχε επιτευχθεί το 2012. Η στατικική αυτή έδωσε σε όλους τους ε, αρμόδιους φορείς ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για δράση ε, που συντόνισε τις προσπάθειες των κατανομελών προς μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική υγείας και ασφάλειας. Επίσης, οι συμβολές από όλους τους ε, πολίτες και τους ε, οργανισμούς, κυρίως και από τις δημόσιες αρχές, οργανώσεις κοινωνικών εταίρων, ε, διαφερόμενους φορείς και πυρογνώμονες του τομέα, ξεκινήσαμε μια διαβούλευση στις 31 Μαΐου 2013, Ταυτόχρονα με τη δημοσίευση της έκθεσης αξιολόγησης. Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε στις 26 Αυγούστου 2013. Πάνω από 500 απαντήσεις λάβαμε. Αυτή τη στιγμή τις αναλύουμε. Και θα δούμε μετά ε, ποια αντίδραση, πώς θα συνεχίσουμε δηλαδή με βάση αυτές τις ε, απαντήσεις. Έχουμε τώρα το ψήφισμα του 2011 για την μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση της νομοδοτήσης για μια νέα στρατηγική που εγκρίθηκε από τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Υγεία και την Ασφάλεια στο χώρο εργασίας και μια επιτροπή ε, που ασχολείται με την, τον αντίκτυπο στην εργασία όλων αυτών των μέτρων. Θα πρέπει βέβαια όλα αυτά να συστηριχτούν με, μια στεναρή βάση αποδείξεων ώστε να εντοπιστεί η ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία, οι προτεραιότητες, οι προκλήσεις και οι προτεραιότητες των επιχειρήσεων. Χρειάστηκε εις βάθος ανάλυση της κατάστασης της υγείας και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας για να εκτιμήσουμε τον αντίκτυπο της στρατηγικής σε διάφορους τομείς, τον αντίκτυπο στους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα της ΜΜΕ και σε σχέση με τα διάφορα εθνικά ε, πλαίσια. Αυτό οδήγησε στον εντοπισμό των βασικών ε, προκλήσεων κατά την περίοδο της προηγούμενης στρατηγικής, όπου θα χρειαστεί να εστιάσουμε περισσότερο την προσοχή μας στο μέλλον. Ταυτόχρονα κάνει η Κομισιόν και μια αξιολόγηση γενικότερα τη ισχύουσα νομοθεσία στον τομέα. Η δημόσια διαβούλευση είχε στόχο τη βελτίωση τη διαφάνεια, τη ε, συμμετοχή του κοινού, που είναι βασικέ αξίε τη ευρωπαϊκή διαδικασία ε, άσκηση πολιτική και για όλου του θεσμού. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Είμαστε τυχεροί γιατί έφτασε η συντάκτρια τη ερώτηση. Απάντησε μεν ο Επίτροπος, έχετε ακούσει τι είπε, θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Περβάνσου Περές για πέντε λεπτά για να παρουσιάσει την ερώτησή της. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Ε, με συγχωρείτε για αυτή τη σύγχυση που επήλθε σχετικά με το ωράριο Ήθελα αυτές τις πληροφορίες μετά τις διαβουλεύσεις ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που κατά κάποιο τρόπο προκαταλαμβάνουν ε, το θέμα που η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ήθελε εδώ να θέσει. Παρ' όλα αυτά, για την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων η μη ανανέωση της στρατηγικής απασχόλησης σχετικά με την υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας είναι πηγή ανησυχίας. Πρώτον, διότι αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αρχή της θητείας της, με την υποστήριξη του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, υιοθέτησε μια στρατηγική 2020, όπου το θέμα του κοινωνικού μοντέλου, της υγείας, της ασφάλειας στον χώρο εργασίας έπρεπε να περιλαμβάνονται στον όλο μηχανισμό. Θυμόμαστε επίσης ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής πέρυσι, εδώ και ένα χρόνο, όταν ανέπτυξε την παρουσίαση για την κατάσταση της Ένωσης, είπε ότι το κοινωνικό μοντέλο ήταν στοιχείο της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για μας το θέμα της υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας είναι στο επίκεντρο αυτού του κοινωνικού μοντέλου. Είναι η καρδιά του κοινωνικού μοντέλου και καμιά φορά έχουμε την εντύπωση ότι επειδή υπάρχει κρίση ενώ η κρίση επιδίνωνε την ανάγκη αυτής της στρατηγική ε, ε, ε, έκανε πιο αναγκαία αυτή τη στρατηγική, απαραμερίστηκε. Δεν αναφέρθηκε αυτό στην προφορική ερώτηση, αλλά ξέρουμε ότι το θέμα μιας νομοθετική πρωτοβουλία στον τομέα των μειοσκελετικών ασθενειών παραμερίστηκε από την ατζέντα προτεραιότητα αυτής τη επιτροπή κατά βάθο το ερώτημα που σας θέσαμε κύριε Επίτροπε είναι να θέλουμε να ξέρουμε γιατί έτσι έχει εξελιχθεί η κατάσταση ενώ αυτή η στρατηγική για την υγεία και η ασφάλεια στο χώρο εργασίας είναι ένα στοιχείο αναγνωρισμένο από όλου ε, τους ενδιαφερόμενους ότι είναι στην καρδιά του κοινωνικού μοντέλου και όχι μόνο είναι ένα στοιχείο ε, προόδου. Γιατί λοιπόν ποια ήταν τα εμπόδια που εμπόδισαν ε, να ανανεωθεί αυτή η στρατηγική. Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων με την προφορική ερώτηση και με την ε, πρόταση ψηφίσματος που θα υποβάλουμε στην Ολομέλεια προσπαθήσαμε να κρατήσουμε το μέτρο και να είμαστε υπεύθυνοι. Δεν θέλουμε να ανοίξουμε πολεμική, θέλουμε να ξέρουμε μέσα στο πλαίσιο που βρισκόμαστε σήμερα, ποια είναι τα εμπόδια που ορθώθηκαν και σας εμπόδισαν εξ ονόματος του σώματος των ε, επιτρόπων να ανανεώσετε αυτήν την στρατηγική που είναι απαραίτητη από την υιοθέτηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 5 Δεκεμβρίου 2011 μιας αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτής της στρατηγικής ασχοληθήκαμε με τον αντίκτυπο αυτής της κρίσης πάνω στους πιο ευάλωτους και εδώ βλέπουμε ότι αυτή η στρατηγική θα ήταν όχι μόνο αναγκαίο να ανανεωθεί, αλλά ότι θα ε, απαντούσε στην ανάγκες που δημιουργούνται και οξύνονται από αυτή την κρίση. Θα έλεγα ότι δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία εμείς ανησυχούμε διότι η κρίση ε, είναι αφορμή, χρησιμεύει ως αφορμή, ως επιχείρημα για να παραμεριστούν αυτά τα μεθεμελιώδη στοιχεία του κοινωνικού μοντέλου ε, στο οποίο είμαστε προσιλωμένοι. Η στρατηγική που είχαμε ε, εκείνη την εποχή είναι μια στρατηγική που πρέπει να ανανεωθεί. Αυτό είναι αλήθεια, διότι οι τεχνολογίες εξελίχθηκαν και λόγω της εξέλιξης των τεχνολογιών νέες δυσκολίες παρουσιάζονται στην υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέτασε το θέμα αυτό, σαφώς το διακύβευμα ε, του στρες στην εργασία που δεν ήταν στην προηγούμενη στρατηγική εμφανίστηκε ως βασικό στοιχείο. Επίσης το θέμα του αντικτύπου αυτής της κρίσης που δυστυχώς γνωρίζει εδώ και πάρα πολύ καιρό η Ευρώπη, εμφανίζεται ως ένα στοιχείο καθοριστικό για την ανανέωση της στρατηγικής. Καταλαβαίνω ότι οι διαβουλεύσεις που είχατε ήταν σημαντικές, χαιρόμαστε αυτό και θέλουμε να προχωρήσετε, αλλά επιτρέψατε μας να πούμε εξ ονόματος Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ότι φοβόμαστε ότι αυτή η στρατηγική θα έρθει πολύ αργά αν έρθει. Και η ελπίδα που είχαμε για το κοινωνικό μοντέλο με την στρατηγική μας έκανε να χάσουμε λίγο χρόνο, να χάσουμε και μπορώ να σας πω εξ ονόματος όλων των μέλων της Επιτροπής λυπούμεθα, θα σας συνοδεύσουμε ε, σε, αν υπάρξει κάποια όθηση για να υπάρξει ένα μήνυμα στο τέλος της θητείας σας, αλλά θέλαμε να έρθει πολύ πιο πριν και θέτουμε την ερώτηση γιατί ποια ήταν τα εμπόδια. Ευχαριστώ. Ακολουθούν οι ομιλητές εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων για δύο λεπτά. Από το ΕΛΚ, ο κύριος Τσάμπα Ωρη. Αγαπητέ Επίτροπε, άκουσα τις απαντήσεις σας με πολύ προσοχή και με ευτυχής γιατί η Κομισιόν δίνει τόση σημασία στην ε, ασφάλεια και στην υγεία στο χώρο εργασίας και στη σχετική στρατηγική. Και εμεί δίνουμε τόσο μεγάλη σημασία σε αυτό το θέμα εδώ στο Κοινοβούλιο, γι' αυτό και έχουμε υιοθετήσει τόσο πολλά ψηφίσματα. Με το τελευταίο τον Ιούλιο, που ο πρόεδρο τη Επιτροπή μα το ανέφερε, αναφέρθηκε και στην μεσοπρόθεσμη έκθεση και συγκεκριμένα ζητήσαμε την Κομισιόν από το 2011, σα θυμίζω, ώστε μέχρι το 2012 θα εξέπαινε η στρατηγική και ότι έπρεπε να ανανεωθεί. Ε, ε αυτό είναι το τέλος της συμβολής μου. Θα μπορούσα να κλείσω γιατί φαίνεται πως η Κομισιόν ε, είχε, ε, την είχε πάρει ο ύπνος γιατί άρχισε τη διαβούλευση με τους κοινωνικού εταίρους αρκετά αργά και ακόμα και τώρα ο Επίτροπος μπορούσε μόνο να μας πει πως οι απαντήσει ήταν γενικά θετικές. Ωραία. Αλλά στην αξιολόγηση και στο σχετικό έγγραφο δεν διαβάσαμε τίποτα για ημερομηνία υποβολής ναι, της νέας στρατηγικής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, γιατί είναι μια αποκλειστική κοινοτική ε, εντολή και αρμοδιότητα. Μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, για ασφάλεια, υγεία. Πολύ σημαντικό θέμα όσον αφορά τον ανταγωνισμό. ευρωπαϊκής οικονομίας. Διαφάνεια και προβλεψιμότητα είναι πολύ σημαντική για τους, ε, τους εργαζόμενους και για τις επιχειρήσεις και είναι προς το συμφέρον των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Αυτό το είδος προθυμίας, διστακτικότητας, καθυστέρησης και αργής προόδου και ακούσαμε και την ε, άποψη της Προέδρου της Επιτροπής μας, δεν είναι κατανοητή και είναι και αντιπαραγωγική προκαλεί κινδύνους για την υγεία, έλλειψη σταθερότητας και αποτελεί σοβαρή απειλή που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Πίτροπε, λοιπόν, γιατί δεν μπορούμε να εγκρίνουμε αυτή τη σημασία. Ποιο είναι το εμπόδιο που σας, που σας ε, κάνει να καθυστερείτε. Ευχαριστούμε. Τώρα για δύο λεπτά επίσης, εξ ονόματος των σοσιαλιστών, το λόγο έχει ο Αλεχάνδρο Θέρκας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Επίτροπε, που ήρθατε μαζί μας τέτοιες ώρες νυχτιάτικα. Και ήθελα να σας πω ότι και για σας και για μας, για την Πρόεδρο και τους συντονιστές, η Επιτροπή μας ανησυχεί βαθύτατα. Το ξέρω κι εσείς. Και συγγνώμη για την αγένεια, Πρόεδρε και Επίτροπε. Ανησυχούμε πολύ ε, γιατί λέτε ωραία λόγια, αλλά τα έργα που είναι στην Ευρωπαϊκή Επίτροπη, η στρατηγική αυτή που ολοκληρώθηκε το 2012, είναι κενή περιεχομένου. Και δεν γνωρίζουμε πολύ καλά γιατί. Γιατί εσείς είπατε ότι γίνανε όλες οι αξιολογήσεις θετικά, όλα πήγαν καλά, όλες οι διαβουλεύσεις είχαν καλή έκβαση. Ε, Προστεί λοιπόν αυτή η ολιγορία και αυτή η καθυστέρηση και δεν μας έχετε δώσει σήμερα ε, σαφή ημερομηνία για το πότε θα εκδοθεί αυτή η στρατηγική. Μήπως επειδή ορισμένοι επιχειρηματικοί κύκλοι λένε ότι τέτοιες ώρες κρίσης δεν μπορούν να επιβαρυνθούν περισσότερες επιχειρήσεις. Μα ακριβώς τώρα ε, στην κρίση έχουμε ατυχήματα εργατικά. Εχθές ήρθαν συνδικαλιστές από ε, τη Γεωργία ε, και είχαν φέτος έξι νεκρούς στην Ισπανία οι Γεωργοί. Αυτά έχουμε να τα δούμε χρόνια αυτά τα εργατικά ατυχήματα και τους θανάτους. Είναι τεράστιες οι κοινωνικές ανάγκες. Μην ακούτε τους επιχειρηματίες που δεν είναι αλληλέγγυοι, ακούστε τους εργαζομένους. Αυξάνεται το άγχος, η κίνδυνη ε, και επιμικρύνεται και ο χρόνος εργασίας. Γι' αυτό κύριε Επίτροπε και κύριε Πρόεδρε, ε, μας λείπουν οδηγίες ε, για ε, τους μεταλλαξιογόνους και καρκινογόνους παράγοντες και άλλα στοιχεία ε, που έχουν μεγάλη σημασία για την υγεία και την ασφάλεια. Σας θυμίζω το άρθρο 31 του Χάρτη των Θεμελιών Δικαιωμάτων και σας λέω ότι υπάρχουν πολλές ερωτήσεις, ακόμα περισσότερες διαβουλεύσεις, αλλά πολύ λίγες απαντήσεις και πολύ λίγες λύσεις. Και τα προβλήματα αντί να λύνονται επιδεινώνονται και σιγά σιγά απομακρύνονται οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι από την Ευρώπη γιατί δεν τη βλέπουν ως σύμμαχο αλλά ως αντίπαλό τους στα θεμελιώδη τους δικαιώματα. Ευχαριστώ εξ ονόματος των φιλελευθέρων για δύο λεπτά η κυρία Χάρκιν παρακαλώ. I want to thank the Commissioner for his answer τον Επίτροπο για τις απαντήσεις του. Χρειαζόμαστε μια τέτοια στρατηγική κατά τη γνώμη μου. Χωρίς στρατηγική τα εθνικά προγράμματα δεν θα μπορούσαν να συνεχίσουν ή να συνεχίσουν με την ίδια ένταση. Πρέπει να έχουμε μια προληπτική κουλτούρα. Αυτή δεν θεωρείται προτεραιότητα. Αυτή η πρόληψη ε, για να προλάβουμε κινδύνους ε, νομίζω θα πρέπει να είναι μέρος της ε, στρατηγικής. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να επανέλθει. Αν δεν υπάρχει νέα στρατηγική δεν θα έχουμε κάτι το ενιαίο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν θα έχουμε προστιθέμενη αξία και η ευρωπαϊκή ε, διάσταση αποκτά λιγότερη σημασία και είναι πάρα πολύ δύσκολο να επαναφέρουμε ορισμένα στοιχεία. Υπάρχει σε εποχή δημοσιονομικών δυσκολιών, πειρασμός να περικόπτουμε πάρα πολλά πράγματα. Βεβαίως αυτό επηρεάζει όλα τα κράτη-μέλη και οι πολίτες είναι απειλούνται ακόμα και περισσότερο. Όσοι εργαζόντουσαν στο Λονδίνο, στον χρηματοπιστωτικό τομέα, είναι ένα παράδειγμα των απειλών, των θυμάτων. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να αλλάξουμε κουλτούρα ε, κυρίως ε, σχέτιμες τις ώρες εργασίας και τις συνθήκες εργασίας. Πού είναι αυτή η κουλτούρα πρόληψης αν δεν έχουμε νέα στρατηγική δεν βοηθάει. Στην Ιρλανδία ε, πριν από το τέλος του μήνα οι νέοι γιατροί θα αρχίσουν απεργίες επειδή δεν, έχουν, δεν υπάρχουν κανονισμοί. Ξέρω ότι δεν μιλάμε για υλοποίηση οδηγίας εδώ αλλά αν δεν έχουμε βοήθεια δεν θα έχουμε την πρόληψη και νομίζω ότι μια νέα στρατηγική θα ήταν μεγάλης βοήθειας. Όπως ε, είπα, ε, οι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερο στρες ε, στην εργασία τους σχετικά με τις ώρες εργασίας ε, και υπάρχουν ε, ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Θα ήταν καλό να είχαμε μια στρατηγική για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Χρειάζεται με τέτοια στρατηγική. Χαιρετίζω την ε, συμφωνία σχετικά με την οδηγία για ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Αλλά έχουμε, βλέπουμε εδώ ότι υπάρχουν εμπόδια. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος των Πρασίνων, για 1,5 λεπτό. Η κυρία Καριμαντελή. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δεκέμβριο του 2011. Το Κοινοβούλιο με μεγάλη πλειοψηφία ψήφιζε τη δική μου έκθεση για αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Υγιεινή και την Ασφάλεια στην Εργασία 2007-2012. Η έκθεση αυτή ήδη έκρουε τον κόδωνα κινδύνου και περιέγραφε την πάρα πολύ ανισχυτική κατάσταση των συνθήκων εργασία στην Ευρώπη. Μερικά στοιχεία μόνο αριθμητικά στην Ευρώπη. Κάθε πέντε δευτερόλεπτα ένα εργαζόμενο ε, είναι θύμα εργατικού ατυχήματο. Κάθε 3,5 λεπτά κάποιο άλλο πεθαίνει από αίτιο που συνδέεται με την εργασία του. Η κρίση δεν μπορεί να είναι πρόφαση ε, για αυτά τα θέματα για να μην ασχολούμαστε και από την έκθεσή μου και μετά συγγύηχθείως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ ανησυχητική νομικό κενό αλλά και πολιτικό πάρα πολύ σοβαρό Ιδού, εδώ και ένα χρόνο το, η Ευρώπη δεν έχει πλέον πολιτικό συντονισμό ως προς την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία για την επόμενη έπτα αιτία. Μας λέγουν και μας εξηγούν και το λέμε και το ακούμε και στους διαδρόμους εφήμες ότι όχι, η γυναίκη ασφάλεια στην εργασία δεν είναι προτεραιότητα. Γιατί, γιατί είναι πανάκριβη. Άκουσον, άκουσον. Εμείς οι οικολόγοι σας το λέμε ξεκάθαρα, πολύ ήρεμα, διαφωνούμε μαζί σας και ήδη από σήμερα απαιτούμε μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία που θα πρέπει οπωσδήποτε να τεθεί σε ισχύ από την 1η 2014. Καθολική ε, κάλυψη ιατροφαρμακευτική ε, για τις μειοσκελετικές παθήσεις, οδηγία από το 2004 για το στρες στην εργασία, όλα αυτά τα λέει η έκθεσή μου πολύ συγκεκριμένα και εγώ τα λέω πολύ ήρεμα. Είναι ηθικό σφάλμα να κλείνουμε τα μάτια ε, σε αυτά τα θέματα, αλλά είναι και οικονομικό σφάλμα, γιατί το κόστος φτάνει μέχρι το 4% του ΑΕΠ, δηλαδή του Ευρωπαϊκού, 500 δισεκατομμύρια για να καλύπτονται αυτά τα εργατικά ατυχήματα. Επίγουσα απάντηση επιβάλλεται γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προστατεύει όλους τους εργαζομένους και να μην χάνουν τη ζωή τους οι εργαζόμενοι προκειμένου να την κερδίζουν. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ε, χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή στρατηγική ε, και προσβλέπουμε και υπολογίζουμε ε, στη δράση σας. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνονται εδώ οι ομιλητές. Με την κυρία Ζούμπερ από το Ιγκούε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Λουξεμβούργο τα τελευταία δύο χρόνια μια κατασκευαστική εταιρεία που αποκαλείται Ασομόδε ε, ε, ε, στην ουσία λειτουργεί και ασκεί δουλεία. Εργάζεται με Πορτογάλους εργαζόμενους που δεν λαμβάνουν ούτε καν τον ελάχιστο μισθό, δουλεύουν σε φρικτές συνθήκες και κοιμούνται σαν τα ζώα όλοι μαζί σε ένα δωμάτιο. Ε, το, εσκα... το σκάνδαλο αυτό δεν είναι μοναδική περίπτωση. Σήμερα με τις πολιτικές προώθησης της ανεργίας, τις τόσο αγαπημένες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να δουλεύουν σε οποιασδήποτε συνθήκες. Τον 21ο αιώνα με συνθήκες του 19ου αιώνα. Βέβαια, οι συνθήκες ε, ασφάλειας και υγείας φυσικά έχουν πάει πίσω λόγω της ε, ύφεση και της ε, κρίσης. Όμως τα στοιχεία σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ανύπαρκτα. Είναι απαραίτητο να λειτουργήσουμε σοβαρά. Γνωρίζουμε ότι πολλές από αυτές τις περιπτώσεις ούτε καν αναφέρονται από τις αρχές, παραμένουν στη σιωπή και στο φόβο. πρόληψη ε, κατάλληλος έλεγχος, ε, δημόσια έρευνα, καταπολέμηση της παράνομης εργασίας που συχνά συνδέεται με απόλυτη απουσία συνθήκων υγείας και ασφάλειας. Η εγκληματικοποίηση αυτών των ε, εμπόρων της εργασίας είναι απαραίτητη γιατί διαρκώς αυξάνεται και θίγεται μάλλον η αξιοπρέπεια των εργαζομένων μας. Σας ευχαριστώ. Τώρα ορισμένοι συνάδελφοι θα λάβουν το λόγο μεμονωμένα και προσωπικά. Η πρώτη κυρία Έντιτ Μπάουερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα ε, να σας πω ότι η ασφάλεια και η υγιεινή συνεργασία είναι πολύ σημαντική, αλλά Υπάρχει και ένα θέμα ανταγωνισμού εδώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετράει την ανταγωνιστικότητα, αλλά δεν έχει στρατηγική για την ασφάλεια και την υγιεινή στην εργασία. Οι στατιστικές επιδεινώνονται, ε, χάνονται θέσεις εργασίας, 53% των εργαζομένων έχουν προβλήματα λόγω ατυχημάτων κατά την εργασία τους. είναι το πιο επικίνδυνο μέρος της καθημερινής ζωής ο χώρος εργασίας. Και αυτό ισχύει και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι συνθήκες εργασίας αλλάζουν, όπως ακούσαμε, λόγω των νέων τεχνολογιών, λόγω της προόδου γενικότερα. Υπάρχουν όμως και άλλοι ε, επιβαρυντικοί παράγοντες. Και όσο ε, παλιώνει και ο εξοπλισμό σε κάποιες επιχειρήσεις, τόσο ε, είναι και πιο επικίνδυνη κατάσταση. Από 216 εκατομμύρια εργαζομένους, 2,5 εκατομμύρια κινδυνεύουν από εργατικά ατυχήματα. Διάβασα σήμερα στις εφημερίδες ότι στη Σλοβακία στη χώρα μας, σήμερα είχαμε ένα μοιραίο εργατικό ατύχημα. Δηλαδή εκατοντάδες πεθαίνουν ακριβώς μετά από εργατικά ατυχήματα. Και κάτι άλλο που τίνουμε να λησμονούμε πολύ συχνά είναι ότι είναι πολύ μεγάλη κίνδυνη. 90.000 άνθρωποι έχουν ε, πάθει εργατικά ατυχήματα χωρίς να χάσουν τη ζωή τους, αλλά παραμένουν ανάπηροι. Υπάρχει η συνθήκη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας και θα πρέπει να μπει ε, στην κοινοτική νομοθεσία, πράγμα που μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει και είναι αποτυχία όλων μας. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει μια νέα στρατηγική για την ασφάλεια και την υγιεινή συνεργασία για να μειωθούν τα αντιχήματα και οι απειλές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Εντίτε Στρέλα για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων είναι προτεραιότητα. Επειδή η Ευρωπαϊκή Στρατηγική εξέπνευσε το 2013, είναι φυσιολογικό να ζητάμε να μάθουμε πότε η Κομισιόν θα παρουσιάσει νέα στρατηγική και ποιοι είναι οι λόγοι αυτής της καθυστέρησης. Το Κοινοβούλιο έχει παίξει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της νομοθεσίας ε, για τις ε, συνθήκες εργασίας που πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στις δυνατότητες και στις ε, ανάγκες των ανθρώπων και όχι τούμπαλιν. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε βελτιώσεις στην νομοθεσία που έχει σχέση με την προστασία των ναι, εγγύων εργαζομένων και των ε, μητέρων που θυλάζουν. Και τον Ιούλιο του 2008 η Κομισιόν παρουσίασε μια πρόταση αναθεώρησης της σχετικής οδηγίας και τον Οκτώβριο του 2010 το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε την εκθεσή μου. Δυστυχώς η υπόθεση αυτή εξακολουθεί να μπλοκάρεται στο Συμβούλιο χωρίς να έχει κάνει κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια η Κομισιόν να έχει ασχίσει κάποιο πίεση ώστε το Συμβούλιο να ξεμπλοκάρει αυτή τη σημαντική έκθεση. Το Κοινοβούλιο επίσης επέμεινε και ήδη αναφέρθηκε από διάφορους ομιλητές αυτό, επέμεινε για την ανάγκη βελτίωσης της νομοθεσίας που σχετίζεται με την προστασία των εργαζομένων απέναντι στις ρευματιπάθειες και τις μυϊκές και σχελετικές παθήσεις. Τα προβλήματα αυτά επηρεάζουν εκατομμύρια ανθρώπους και αποτελούν μεγάλο βάρος για το σύστημα υγείας και το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 25% των ε, μεγάλων μακροχρόνων αποσιών προκύπτουν από και οφείλονται σε ρευματικές παθήσεις και παθήσεις μυϊκές ή σκελετικές. Εγώ ασχολούμαι με αυτή την ομάδα ε, στο Κοινοβούλιο και τις σχετικές παθήσεις αυτές που σας αναφέρω. Είναι λοιπόν προφανές, ε, κύριε Επίτροπο, ότι χρειαζόμαστε μια νέα στρατηγική που να είναι προσαρμοσμένη στις νέες πραγματικότητες και στην εξέλιξη της κοινωνίας μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Εντίτ. Για δύο λεπτά επίση, το λόγο τώρα έχει η κυρία Γιαζοβιέτσκα. Ευχαριστώ πολύ. Μετά πολλές αλλαγές συνθήκων η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάντοτε την αρμοδιότητα που μοιράζεται με τα κράτη-μέλη σχετικά με την απασχόληση και την υγεία και πολλά κράτη-μέλη είναι επιφυλακτικά να υιοθετήσουν ε, κανόνες πιο προχωρημένους στον τομέα αυτό. Νομίζω ότι το θέμα της υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας αποδεικνύει ότι οι δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο από το 1978 είναι ε, επιθυμητές και αυτό έχει επιτευχθεί με μέσα μη ε, δεσμευτικά και η στρατηγική που υιοθετήθηκε επέτρεψε την βελτίωση της ισχύουσας νομοθεσίας. Νομίζω ότι στα επόμενα χρόνια απαιτούνται εργασίες και πρόδι ε, και εκπλήσωμε διότι η Κομισιόν αργεί να παρουσιάσει μια νέα στρατηγική. Οι δράσεις για την βελτίωση της υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας είναι απαραίτητες για να επιτύχουμε τους στόχους που θέσαμε για το 2020. Λόγω ε, της ε, τάσης γύρανσης ε, του πληθυσμού ε, και της παράτασης της επαγγελματικής ενασχόλησης του πληθυσμού πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υιοθετήσουμε μέτρα που να επιτρέπουν να προσαρμόσουμε τις θέσεις εργασίας σε άτομα άνω των 55 ετών. Θα πρέπει επίσης να έχουμε δράσεις προληπτικές σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και την υγεία των εργαζομένων και θα πρέπει να ασχοληθούμε με τους νέους, με ειδικέ δράσεις, πράγμα που θα επέτρεπε να βελτιώσουμε την επαγγελματική τους κινητικότητα. Υπάρχουν επίσης τεχνολογικές αλλαγές που εμφανίζονται σύντομα που επηρεάζουν την υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραδέχθηκε πάρα πολλές φορές ότι η στρατηγική 2007-2012 είχε θετικά αποτελέσματα παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ότι υπάρχουν τομείς που, όπου υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, γιατί δεν υπάρχει νέα στρατηγική για τα 2013-2020 όπως είχε αναγγελθεί. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ και εγώ. Τελευταία ομιλήτρια στη συζήτηση αυτή είναι η κυρία Κώστελο. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και Επίτροπε, σας ευχαριστώ που είστε απόψε εδώ. Εγώ συμμερίζομαι την ανησυχία του συναδέλφων όσον αφορά την απασχόληση, την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων για την καθυστέρηση της νέας στρατηγικής για την υγεία και την ασφάλεια. 5.000 θάνατοι στο χώρο εργασίας ετησίως και φέτος στην Ιρλανδία σκοτώθηκαν και δύο παιδιά. Ε, χρειάζεται οπωσδήποτε νέα στρατηγική υγείας και ασφάλειας. Με αυτό το ρυθμό δεν θα έχουμε νέα στρατηγική μέχρι το 2014 και η στέρηση αυτή είναι απαράδεκτη. Ιδιαίτερα αν δει κανεί του λόγου για του οποίου χρειαζόμαστε αυτή τη στρατηγική. Αυξημένη χρήση χημικών, γύραση του εργατικού δυναμικού, μειοσκελετικέ παθήσει, ε, καρκίνοι που σχετίζονται με την ε, εργασία, στρε. Ε, πρέπει όλα αυτά να αντιμετωπιστούν. Η υγεία και η ασφάλεια είναι καλή, είναι σημαντική για του εργαζόμενου και όπω υπόθηκε προστατεύει και το κοινωνικό μοντέλο αλλά είναι καλύτερο και για τις επιχειρήσεις, γιατί καλύτερη υγεία και ασφάλεια συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση της εταιρεία, στην ευημερία του προσωπικού, στην απόδοση και στην ικανοποίηση από τη δουλειά. Αντί να κατηγορούμε την κρίση, και να χρησιμοποιούμε την κρίση ως, ευκαι... Ε, ε, δικαιολογία για να μην εφαρμόζουμε αυτή τη στρατηγική. Αντιθέτως, χρειαζόμαστε μια στρατηγική που θα, είναι... θα ανταποκρίνεται στον 21ο αιώνα και θα μας βοηθήσει. Η καθυστέρηση έχει διαρκέσει αρκετά. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει τις ευθύνες της και να προτείνει νέα στρατηγική. Ευχαριστώ, Εμέρ. Συγγνώμη. Ακούστε με. Θέλετε να κάνετε ερώτηση στην κυρία Έμερ Κώστελο. Αυτό ζητάτε. Όχι. Στο Κατσιάι ζητάτε το λόγο. Θέλετε να εγγραφείτε στη διαδικασία Κατσιάι. Η γαλάζια κάρτα είναι για, συζήτηση, για ερώτηση στην κυρία Κοστέλο. No, entonces, entonces... Εντάξει. Είναι η συνάδελφος από την Κροατία και μπράβο της που κάθισε τόσο αργά. Απλώς ήθελα να σας πω ότι χρειάζεται για το CATCI λευκή κάρτα, όχι γαλάζια. Ε, λευκή κάρτα για να γραφτείτε στη διαδικασία του CATCI. Εντάξει, ωραία. Ναι, ναι, βεβαίως και φυσικά θα σας δώσουμε το λόγο, λίμωνο. Ξέρετε ότι έχετε ένα λεπτό για την παρέμβασή σας και σας συγχαίρω για το ενδιαφέρον σα για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ζητώ συγγνώμη για τη σύγχυση. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, λιγότερο από 4 εκατομμύρια Ευρωπαίων, μάλλον περίπου 4 εκατομμύρια, ε, τραυματίζονται στην εργασία και 5.000 χάνουν τη ζωή τους. Ε, είναι σοβαρά αυτά τα στοιχεία ε, και οφείλονται σε κάποιους εργοδότες που αγνοούν και παραγνωρίζουν κάθε κανόνα προστασίας των εργαζομένων. Ε, αλλά και οι ίδιοι εργαζόμενοι δεν έχουν επίγνωση της σημασίας ε, να προστατεύουν την υγεία τους κατά την εργασία. Η πρόληψη είναι βασικό στοιχείο και θα πρέπει να ποντάρουμε εκεί. Θα πρέπει να προστατεύουμε την υγεία και τη ζωή των εργαζομένων μας. Προφανώς υπάρχουν και οικονομικές επιπτώσεις και συνέπειες. Κάθε εργαζομενός στην Κροατία ε, παίρνει 10 μέρες άδεια ε, για ε, θέματα υγείας, αναρωτική δηλαδή, ε, που σημαίνει 110.000 ώρες το χρόνο, με οικονομικές συνέπειες όπως σας είπα. Θα πρέπει αυτή η στρατηγική να επιταχυνθεί στην έγκρισή της και να υπάρχει ενιαία ευρωπαϊκή προσέγγιση το συντομότερο. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι. Πριν δώσω το λόγο στον Επίτροπο για να κλείσει, θα ήθελα να τονίσω κάτι που με ενδιαφέρει να εγγραφεί στα πρακτικά. Κοιτάξτε, 11 παρεμβάσεις είχαμε. Από τις 11 παρεμβάσεις, οι 9 ήταν γυναίκες και θέλω να το τονίσω. Αυτό δεν είναι ίσονο σημασία, είναι άξιο πρόσεκτο. Τι έγινε, δεν έχετε γαλλική διερμηνία. Λοιπόν, έλεγα, από τις 11 παρεμβάσεις, οι 9 που μίλησαν ήταν γυναίκες. Είναι πραγματικά αξιοσημείωτο. Εγώ συμπεράσματα δεν βγάζω. Ε, ελπίζω να τα βγάλουμε όλοι μας. Και μάλιστα υπήρξε και άλλη συνάδελφος ε, που δεν πήρε το λόγο. Δύο άντρες μίλησαν, εκτός από τον Επίτροπο και εμένα που βρισκόμαστε εδώ γιατί είναι υποχρέωσή μας. Αλλά συμμετοχή στη συζήτηση είναι πραγματικά άξιο σημείωτο και θέλω να εγγραφεί στα πρακτικά για να παραμείνει. Διότι είναι πραγματικά σημαντικό. Από τους 11, 9 γυναίκες και 2 άντρες για ένα θέμα με τέτοια εμβέλεια και τέτοια κοινωνική σημασία. Κύριε Πίτροπε, έχετε το λόγο για να ολοκληρώσετε τη συζήτηση. Παρακαλώ. Uh, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ όσους συμμετείχαν στη συζήτηση και την κυρία Μπέρες η οποία έθεσε ε, το ερώτημα για την υγεία και ασφάλεια. Θα ήθελα να τοποθετήσω το θέμα σε ευρύτερο πλαίσιο για να κατασταθεί σαφές για όλους ότι ότι έχουμε μεγάλες ζημιές ως προς τον αριθμό των θέσεων εργασίας και την επιδείνωση των συνθήκων εργασίας και θα πρέπει να επιταχύνουμε την εργασία για να περιλάβουμε τις συνθήκες εργασίας για όλες τις ε, κατηγορίες εργαζομένων. Ε, πρόσφατα η Επιτροπή βρίσκεται, ε, βρέθηκε σε συνεχή διάλογο με όλους τους ενδιαφερόμενους για την οικία και ασφάλεια, όχι μόνο για την ε, πρόοδο που έγινε σε ειδικού φακέλους ε, όπως η έκθεση σε υλομαγνητικά πεδία. Είχαμε υποστήριξη γενική όλων των κομμάτων για την υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας και κυρίως από τις πολιτικές ομάδες που αντιπροσωπεύτηκαν σήμερα στη συζήτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χαιρετίζουμε το γεγονός αυτό και χωρίς αυτήν την υποστήριξη όλων δεν θα είχαμε την ευκαιρία να επιτελέσουμε πρόοδο. Ο κύριος Έριπ και η κυρία Μπάουερ ε, αναφέρθηκαν στεναρά ε, στο θέμα ότι είναι επίσης θέμα ενιαίας αγοράς. Ε, το θέμα των ίσων όρων, ε, του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά καθιστά αναγκαίο να έχουμε το θέμα αυτό ως τομέα πολιτικής αρκετά σημαντικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά θα ήθελα να τονίσω δύο άλλες απόψεις δεν είναι μόνο η εξωτερική διάσταση. Τα πρόσφατα χρόνια θα μάθατε ότι εγώ εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετείχα σε σημαντικό ε, διάλογο ε, για, ε, για, για τις αναδυόμενες χώρες. Τα ατυχήματα που είχαμε στο Μπαγκλαντές απαιτούν ε, συνεκτικές απαντήσεις από τις πιο ανεπτυγμένες χώρες και κυρίως την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και έχουμε απόκριση στην διεθνή κοινότητα σχετικά με αυτό το σημαντικό ατύχημα. Είναι σημαντικό να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαφυλάξει την αξιοπιστία της μόνο αν εξακολουθήσει να δρά στεναρά και συνεκτικά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και, αν, για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στην ενία αγορά. Νομίζω ότι η κυρία Κοστέλο ανέφερε ένα κάτι το σημαντικό που είναι η σύνδεση ανάμεσα στην υγεία και η ασφάλεια και τις δημογραφικές αλλαγές. Έχουμε μια εργατικό δυναμικό στην Ευρώπη που συρρυκνώνεται ε, και που γυράσκει και για να παραμείνει το το δυναμικό αυτό το εργατικό ε, ανταγωνιστικό και να συμβάλλει σε ευημερία στην επόμενη δεκαετία θα πρέπει να επενδύσουμε στην υγεία και ασφάλεια διότι θα αποδώσει αυτό σχετικά με, με, με θέματα όπως οι μειοσκελετικές ε, διαταραχές ε, δεν χρειάζεται να σας πω περισσότερα και σύμφωνο ότι η κρίση δεν πρέπει να αποτελεί πρόφαση ούτε ε, να έχουμε ε, βραχυπρόθεσμη ενόραση, θα πρέπει να βλέπουμε μακρυπρόθεσμα πώς μπορούμε να ωφεληθούμε από αυτές τις πολιτικές. Αλλά το ε, ερώτημα κλειδί όταν θεωρούμε μια νέα στρατηγική και τον χρονισμό της είναι η προστιθέμενη αξία ενώ τα κράτη-μέλη κάνουν προόδους όπως την έκθεση, παρόντος χάρη στο κάπνισμα, εκεί υπάρχει πρόοδος στο επίπεδο των κρατών μελών. Επίσης έχουμε μια ε, εξέλιξη στις καλές πρακτικές ε, των εταιριών, διότι ξέρουν οι εταιρείε αυτό που τόνισε η κυρία Χάρκιν, ότι η υγεία και η ασφάλεια στο χώρο εργασίας δεν είναι μόνο μια δαπάνη, αλλά και μια επένδυση. Επίσης ε, έχουμε ένα σημαντικό έργο για να υλοποιήσουμε, να εφαρμόσουμε την υφιστάμενη νομοθεσία που υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι σημαντικό έργο σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία και την κληρονομιά της στρατηγικής του παρελθόντος. Προσωπικά δεν έχω καμία αμφιβολία για τη σημασία των μελλοντικών δράσεων στον τομέα αυτό. Σήμερα το πρωί ο πρόεδρος Μπαρόζο τόνισε την σημασία της στρατηγικής 2020 για τις μελλοντικέ δράσεις της Κομισιόν και αυτή η στρατηγική όπως γνωρίζετε έχει αριθμητικούς στόχους σχετικά με το ρυθμό απασχόλησης να αυξηθεί στο 75%. Νομίζω ότι μια καλή πολιτική ευρωπαϊκή στον τομέα της υγείας και ασφάλειας μπορεί να συμβάλλει στο στόχο αυτό και να αποτελέσει σημαντικό ε, μέρος ε, της προσπάθειας για να έχουμε το 70% απασχόλησης. Ε, οι χώρες που έχουν 75% είναι αυτές που έχουν τις καλύτερες πρακτικές ως προς την υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Ο κύριος Μπαρόζο επεσήμανε την έλλειψη αποφασιστικότητας ως μεγάλο κίνδυνο που απειλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα αυτό που μπορώ να σας πω ότι η έλλειψη αποφασιστικότητας επίσης παίζει μεγάλη σημασία στον τομέα αυτό αλλά με δυνατή στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μπορέσουμε ίσως να υπερνικήσουμε αυτό το εμπόδιο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Λάβαμε μία πρόταση ψηφίσματος για να κλείσει αυτή η συζήτηση και ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση. Αύριο θα γίνει η ψηφοφορία στις 12 το μεσημέρι. Θα ήθελα οπωσδήποτε να ευχαριστήσω και να συγχαρώ όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτή τη συζήτηση, πολύ ενδιαφέρουσα.